Η περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διακόπηκε στι 14 Απριλίου συνεχίζεται. Αγαπητοί συνάδελφοι. οι περισσότεροι ξέρουν ακριβώς τι έγινε στις 29 ε, Απριλίου 1986. Είναι στη μνήμη μας πριν από 30 χρόνια κυρίες και κύριοι, στις 26 Απριλίου 1986